Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε ένα διορθωτικό σε ένα κείμενο που εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του κανονισμού αν δεν διαφωνήσει ή προπάλλη ένσταση μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται. Το κείμενο θα το βρείτε στο Seance on Direct και θα δημοσιευθεί και ο τίτλος στα πρακτικά της παρούς συνεδρίασης. Σύμφωνα με το άρθρο 74 ε, του κανονισμού, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω ε, τα κείμενα που